Σας αναφέρω ότι υποδεχόμαστε σήμερα μια αντιπροσωπεία βουλευτών και άλλων επισκεφτών από την πολιτεία των μεγάλων ουραλίων από τη Μογγολία και επίσης καλεσμένους από την αποστολή της Μογγολίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βρίσκονται στα επίσημα θεωρία. Τα μέλη της αντιπροσωπείας είναι στις Βρυξέλλες για να συναντηθούν με τους ομολόγους του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 7η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μογγολίας. Αυτό θα ενισχύσει την, ε, ε τη σχέση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Μογγολίας που είναι αυξανόμενη σημασία. Οι επισκέπτε επίση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από πρώτο χέρι την εργασία του Κοινοβουλίου μας και θέλω να ευχηθώ καλή διαμονή στην αντιπροσωπή αυτή στην ε, διάρκεια της επισκέψης του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση της κυρίας Ατ Γουλ για την κοινωνική δράση σε σχέση με την φαλαινοθή.